η έκθεση της ε, Λιλιάνα Ροτρούγκες για την ενδυνάμιση των κοριτσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της εκπαίδευσης. Η εισηγήτρια έχει το λόγο παρακαλώ για τέσσερα λεπτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη τα οποία συνεισέφεραν σε αυτήν την έκθεση. Ε, με βοήθησαν πάρα πολύ συνεισφορές σας. Ε, καταλήξαμε σε συμβιβασμούς και αυτό ήταν νομίζω η νίκη. Ε, είναι πολύ σημαντικό τα κορίτσια να μπουν στο επίκεντρο της δράσης μας. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα εγγυηθούμε ότι στο μέλλον όλοι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τρόπο πραγματικά αποτελεσματικό και όχι μόνο στα λόγια. Ορισμένοι θα πούν ότι η κατάσταση είναι καλύτερη σε σχέση με πριν από μερικά χρόνια. Η αλήθεια είναι αυτή, πράγματι. Η κατάσταση είναι καλύτερη, αλλά τα πράγματα ε, βελτιώνονται πολύ αργά, ακόμα και μέσα στα ευρωπαϊκά όργανα. Οι γυναίκες πολύ συχνά εξακολουθούν να ζουν ε, διάκρισης βάρος τους. Είναι πολύ σημαντικό να καταργήσουμε προκαταλήψεις και στερεότυπα. Και αυτό πρέπει να γίνει από την παιδική ηλικία. Ε, αγόρια, κορίτσια, άντρες και γυναίκες μπορούν να αλλάξουν την κοινωνική δομή. Αυτή η έκθεση συμπίπτει με την Διεθνή Μέρα της Γυναίκας ε, που έχει θέσει ε, την εκπαίδευση της γυναίκας ως εργαλείο άσκησης εξουσίας. Οι, οι γυναίκες θα, μάλλον τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ε, την ε, σχολική, το ότι η σχολική κουλτούρα θα ε, συνάδει με τους στόχους μας. Τα σχολικά προγράμματα θα πρέπει να προσαρμοστούν. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αποφύγουμε τις διακρίσεις από τη μικρή ηλικία των παιδιών. Είναι πολύ βασικό αυτό για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ε, ελευθερία, ισότητα και αδελφότητα θα πρέπει να είναι το, στο πνεύμα μας. Δύο βασικοί στόχοι. Πρώτον, να εξασφαλίσουμε την ισότητα των κορισιών μέσω της εκπαίδευσης. Δεύτερον, ε, να εφαρμόσουμε τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη των διακρίσεων με βάση το φύλλο. Πέντε ειδικοί στόχοι. Ε, σχολική κουλτούρα ισότητας των φύλων. να παρακολουθούμε κριτικά τα προξιολικά προγράμματα, να εξασφαλίσουμε την ισότητα των δύο φύλων σε ό,τι αφορά την λήψη προσωπικών και επαγγελματικών αποφάσεων, να βελτιώσουμε την ε, παρουσία των γυναικών σε υψηλέ θέσει, να προωθήσουμε την ισότητα σε ό,τι αφορά την οικονομική ανεξαρτησία. Αυτή είναι η πέντε ειδική στόχη. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτούς τους στόχους. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες ιδεολογικέ διαφορές. Ε, αρνούμαστε σε αυτή την έκθεση ε, ότι ε, υπάρχουν κάποιοι οποίοι εξουσιάζουν και κάποιοι οποίοι εξουσιάζονται. Παρόλο ότι πρόκειται για μια έκθεση για την ενδυνάμωση των κοριτσιών, είναι σαφές σε όλους μας ότι οι άντρε και τα αγόρια είναι απολύτως απαραίτητο να συμμετάσχουν γιατί αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Οι, τα κορίτσια θα πρέπει να προστατευθούν με τη συμμετοχή και την προσπάθεια όλων. Ελπίζω ότι θα υπερψηφιστεί αυτή η έκθεση. Η λογική είναι να προστατεύσουμε τα κορίτσια μας που σε λίγο θα γίνουν γυναίκες. Προστατεύοντας τα κορίτσια είναι σαν να προστατεύουμε τις γυναίκες και το μέλλον της Ευρώπης. Ε, ευχαριστώ. Και τώρα διαδικασία Κατστιάη. Κυρία Πέτρη. ένα λεπτό. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ο στόχος της εκθέσεως είναι η ανατροπή των παραδοσιακών εικόνων της οικογένειας και της κοινωνίας και δεν μπορώ να την υποστηρίξω. Πρέπει βεβαίω να βελτιωθεί η πρόσβαση των κοριτσιών στην εκπαίδευση, αλλά από τον έβηχο αυτό τίτλο κρύβονται άλλα πράγματα. Η έκθεση φτάνει μέχρι και στην αναφορά της ε, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης μέσα από το σχολείο. Αυτό αντίκειται σε κάθε νέα δικαίου. Οι γονείς, και αυτό το λένε οι διεθνείς συμβάσεις, είναι οι πρώτοι που διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους. Αυτό αποτελεί λοιπόν παραβίαση της ε, οικογένειας, δεν έχει καμία σχέση με την εκπαίδευση και μόνο στόχο έχει την ανατροπή της οικογένειας και της εικόνας της κοινωνίας μας. Γι' αυτό δεν μπορώ να υποστηρίξω αυτήν την εκθέση. Ο κύριος Σάντος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει ως καθήκον την πρόθεση της ισότητας των δύο φύλων. Όλα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν ε, πρόσβαση σε μια δημόσια εκπαίδευση δωρεάν και χωρίς διακρίσεις. θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προστασία της ισότητας των δύο φύλων. Ο, αυτό προτείνει η συγκήτρια, ε, είναι, σημαίνει ότι η δημοκρατικοποίηση της ε, παιδείας θα οδηγήσει στην ε, ισότητα των δύο φύλων και στην εξάλληψη των διαφορών οικονομικών και κοινωνικών. Η ενδυνάμωση των κοριτσιών θα σημαίνει η ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι πεπισμένο ότι η ανάπτυξη της προσωπικότητας, ε, η ανεκτικότητα, ε, η υπευθυνότητα και η ελεγγύη θα βελτιώσει ε, την κοινωνική κατάσταση όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στηρίζω αυτή την έκθεση της κυρίας Ροντρίγκες. Ο κ. Μαριάς έχει το λόγο τώρα. Για ένα λεπτό. κύριε Πρόεδρε. Η ενδυνάμωση των κοριτσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω τη εκπαίδευση είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμβάλλουν στον εκδημοκρατισμό τη εκπαίδευση, ώστε να διασφαλιστεί ότι προωθείται έτσι η ισότητα των δύο φύλων και δίνει σε άνδρες και γυναίκες ίσες ευκαιρίες για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη επιπλέον θα πρέπει να οργανωθούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης πάνω στις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και να βελτιωθούν οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις και στην αγορά εργασίας. σε όλα τα προγράμματα διδασκαλίας θα πρέπει να συμπεριληφθεί η διαπαιδαγώγηση όσον αφορά τα δικαιώματα των δύο φύλων. οποιαδήποτε πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης πάνω στο θέμα της διάκρισης των δύο φύλων θα πρέπει να ενισχύεται μέσω της εκπαίδευσης θα πρέπει να καταρριφθούν τα στερεότυπα που αφορούν τα δύο φύλλα και να προωθηθούν οι γυναίκες σε όλους τους χώρους εργασίας ώστε να ενδυναμωθεί έτσι και η κοινωνία γενικότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαραγκάλ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διάλογος και καλή δουλειά μας οδηγεί σε καλό αποτέλεσμα και από την Επιτροπή Γυναικών, ε, την κυρία Ροντρίγκε, αλλά και από την Επιτροπή Πολιτισμού. Εργαστήκαμε, νομίζω, προς τη σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, ποτέ δεν ολοκληρώνεται η εργασία για την ισότητα των φύλων, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να έχουμε χειραφέτηση στον τομέα της εκπαίδευσης εάν θέλουμε να έχουμε οποιαδήποτε δυνατότητα στην προηγούμενη έκθεση, πρέπει να υποστηρίξουμε όλοι με ενθουσιασμό ε, την έκθεση της κυρίας Ροντρίγκες. Αλλιώς ε, απατώ, ε, αυταπατώμαστε όλοι. Δεν ήθελα να λάβω το λόγο σε αυτή τη συζήτηση, αλλά είδα κάποιες επιθετικές συμπεριφορές για την οικογένεια, για την Ευρώπη και αντιλήφθηκα αυτό το οποίο συμβαίνει στην πραγματικότητα. Η έκθεση αυτή είναι απόδειξη της κατεπίγουσας ανάγκης να προχωρήσουμε στο δρόμο που μας προτείνεται για την ισότητα των φύλων, για την καταπολέμηση των στερεοτύπων και το καθεξής. Σας ε, επιβεβαιώνω σήμερα ότι θα συμφωνήσω με την κυρία Ροντρίγκε και τους υπόλοιπους συναδέλφους για τα όσα ε, έκαναν. Θα πρέπει να υπάρχει μια ισότητα που θα σέβεται και τη διαφορετικότητα. Θα πρέπει όλα αυτά να ξεκινήσουν από το σχολικό περιβάλλον για να μπορέσουν στη συνέχεια να έχουν όλοι τη σταδιοδρομία που τους αξίζει και να είναι κύριοι του εαυτού τους. Η κυρία Ζαμπόρσκα τώρα, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Είμαι κατά της, ε, του δικαιώματος ε, των ε, γονέων να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους όπως επιθυμούν. Είναι φιλόδοξο το πρόγραμμα αυτής της έκθεσης. Ε, ε, Ζητά η συγγήτρια και πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα είναι παραβίαση των συνθήκων. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ε, απαιτεί έγκριση νομοθεσίας για την παιδεία και το ποινικό δίκαιο. Αλλά βάσει Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την εξουσιοδότηση να εγκρίνει τέτοια νομοθεσία. Ήδη υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και επιβεβαιώθηκε στο παρελθόν ότι η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα είναι ε, ασύμβατη ε, με τις ευρωπαϊκές εκθέσεις. Γι' αυτόν λοιπόν και για διάφορους άλλους, ε, ευρωπαϊκές συνθήκες, συγγνώμη, γι' αυτόν και για διάφορους άλλους λόγους είμαστε κατά της έκθεσης και θα την καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής από τη Σλοβακία, ο κ. Κρίτεκ. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, ούτε εγώ θα ευχαριστώ τον κύριο Ροτρίγκης για την έκθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε προσφέρει μεγάλη ελπίδα στους Σλοβάκους για δημοκρατία και πλουραλισμό. Πού είναι όμως η δημοκρατία δέκα χρόνια μετά. Βλέπουμε να ξεπερνούνται τα όρια των αρμοδιοτήτων και της επικουρικότητας η πολιτική για το φύλλο δεν μπορεί να οριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να ακούσουμε τις φωνές των πολιτών της Ευρώπης, της Σλοβακίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και να μην παραβιάσουμε τα δικαιώματα αυτά. Η έκθεση Φερέρα, η έκθεση Ροτρίκες αποτελούν αποδείξεις ότι παραβιάζονται οι βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εθνική κυριαρχία των κρατών μελών δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Γκαρίκα, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μεγάλο θέατρο από τα αριστερά του ημικυκλίου, αλλά Μόνο θέατρο, χωρίς ουσία. Εγώ θα το καταψηφίσω λοιπόν. Η πολιτική της εκπαίδευσης δεν είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον οδηγό σπουδών των παιδιών μου και δεν υπάρχει κανένας λόγος τα παιδιά μου να μαθαίνουν ε, ότι υπάρχουν διεμφυλικοί μια γυναίκα που μόνη να τρέφει τα παιδιά της, ένας πατέρας μόνος του, ίσως θα μπορέσει καλύτερα να εξηγήσει τη ζωή στα παιδιά παρά μια ομάδα που θα επιβάλλει στα σχολικά εγχειρίδια αυτές τις ιδέες. Και θέλω να πω ότι η Ευρώπη έχει πολλά προβλήματα. Δεν χρειάζεται ε, σεξουαλική αγωγή στην Ευρώπη, στα σχολεία, ίδια για όλα τα σχολεία. Α σταματήσουν λοιπόν αυτέ οι εκθέσει πρωτοβουλία γιατί αρχίζουν και μα ενοχλούν πια. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκέρικε, ήσταν και ο τελευταίος ομιλητής εκ μέρους του Κοινοβουλίου. Τελευταίος όμως και εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, Επίτροπος Τίμπορ Ναύρατσισκ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Επιτροπή καλωσορίζει την έκθεση «Ενδυνάμωση των κοριτσιών και γυναικών μέσω της εκπαίδευσης», η οποία τονίζει πως η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι κρίσιμη σημασίας και το πρακτικό παράδειγμα είναι κρίσιμη σημασίας για να αντιμετωπίσουν τις ανισότητες μεταξύ των φύλων ε, τα κορίτσια και οι γυναίκες σε πρώιμο στάδιο και σε μικρή ηλικία. Έχουμε να κάνουμε σημαντικά επιτεύγματα, μεγαλύτερη αναγνώριση της ισότητας των φίλων ως αντικείμενο εκπαίδευσης. Οι γυναίκες έχουν ενισχύσει τη συμμετοχή τους στην, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. συμμετέχουν ε, και σε διάφορους τομείς ε, μελέτης, ε, σε κατηγορίες σπουδών που παλαιότερα θεωρούνταν μονοπόλιο των ανδρών. Επίσης, Βλέπουμε σημαντικές αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα. Μπορεί οι γυναίκες να έχουν υψηλότερα πτυχία, ωστόσο παραμένει η υποεκπροσωπούμενο το γυναικείο φύλλο στις επιστήμες των μαθηματικών, της φυσικής, στις στερεοδρομίες που έχουν να κάνουν με την έρευνα και την ε, τεχνολογία. Δεν αναγνωρίζονται οι, τα επιτεύγματα τους και ενώ είναι περισσότερες οι γυναίκες πτυχιούχοι έχουν καλύτερες επαγγελματικές επιτυχίες οι άνδρες με, μια διαφορά κατά 4% μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο ανισότητες. Επίσης υπάρχουν και στον ε, χώρο των διδασκάλων όπως και στον, ε, στα στελέχη. Στα σχολεία, τα πανεπιστήμια, δάσκαλοι δεν καλύπτονται ακόμα από τις πολιτικές για την ισότητα των φύλων. Η διάσταση, των οποίων καταγράψει, η διάσταση της οποίας καταγράφεται στην ε, στρατηγική για την ισότητα τον προηγούμενο Μάρτιο και ύστερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία και τη Δανία συναντήθηκαν οι Υπουργοί Εκπαιδείας στη Γαλλία στο Παρίσι για να προαγάγουν τις πολιτικές της κατάρτισης και της εκπαίδευσης χωρίς διακρίσεις και χωρίς φανατισμούς. Μια από τις κύριες αξίες μας, μια από τις αξίες που οι Ευρωπαίοι Υπουργοί αναλαμβάνουν να προαγάγουν. Το Erasmus Plus επίσης είναι το πρόγραμμα χρηματοδότησης που προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για δουλειά σχετική με την ισότητα των φύλων. Η ισότητα των φύλων πρέπει να ξεπεράσει λοιπόν τις πολιτικές προθέσεις και να, να μετατραπεί σε πραγματικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στους δασκάλους, η στάση των οποίων μπορεί να διευκολύνει την αλλαγή συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την ισότητα των φίλων μας, των πολιτικών και των προγραμμάτων μας που καταγράφουν νέες προτεραιότητες ε, σε στην συνεργασία με τα κράτη-μέλη και στο στατικό πλαίσιο γιατί το 2020 ταχύτερη πρόοδος είναι δυνατή. Μπορούμε να, πρέπει να προχωρήσουμε από τον εντοπισμό των ε, προβλημάτων στις λύσεις, να δώσουμε πόρους ε, με στοιχεία, με μετρήσιμους στόχους και παρακολούθηση της πρόοδου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να υλοποιηθεί στην πράξη αυτή η έκθεση σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Thank uh, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επιτροπέ.